Δεν θα ξεκινήσουμε αμέσως αγαπητοί συνάδελφοι γιατί περιμένουμε τον Πρόεδρο ο οποίος πρέπει να κάνει μια τραγική ανακοίνωση δυστυχώς και πρέπει να σας ζητήσω να περιμένετε ε, λίγα λεπτά ακόμα.